Στι στις 8.30 μέχρι τις 2 η συνεδρίαση και από τις 3 μετά μέχρι τις 4. Έχετε την ε, ημερήσια διάσταση.